επόμενο θέμα έχω δύο ανακοινώσει. Δεν υπήρξε καμία αντίρρηση εντό 24 για τι προτάσει Επιτροπή Γιούρι που ανακοινώθηκαν ε, κατά την ανακήρυξη τη Αναξολομέλεια σε σχέση με δύο κατεξοδότηση πράξεων. Κατ' εφαρμογή λοιπόν του άρθρου 105 παραγράφου 6 θεωρούνται εγκεκριμένε αυτέ οι συστάσει και θα δημοσιοποιηθούν με τα εγκεκριμένα κείμενα αύριο την Τετάρτη 5 Ιουλίου